για έξι ψηφίσματα για τη Γουινέα και θα δώσω το λόγο στους συντάκτες. Πρώτα στην κυρία Ντεκεζέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον αυτού του ζητήματος ξεπερνά κατά μεγάλο βαθμό την προσέλευση των βουλευτών, την πολυπληθή προσέλευση των βουλευτών. Εκφράζω και πάλι την λύπη μου και για τη δική μου ομάδα και για του υπόλοιπου. Η Γουινέα Κονακρή χρειάζεται την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Μετά από την, ε, το θάνατο του πρώτου Κοντέ, ένας νέος στρατιωτικό πήρε την εξουσία. Είχε υποστήριξη στο εσωτερικό, παρά το γεγονός ότι στο εξωτερικό δεν είχε μεγάλη υποστήριξη, υποσχόμενος ελεύθερες εκλογές και μια πολιτική κυβέρνηση στο μέλλον. Και μετά από την ε, ολέθρια διαχείριση της προηγούμενης κυβέρνησης που δεν μπόρεσε να δώσει ούτε καν τις ε, βασικές υπηρεσίες στους πολίτες, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Η εκλογική εκστρατεία λοιπόν του πρώην Προέδρου βασίζεται σε όλους τους πόρους της πόλης της ε, Γουινέας Κονακρή. Αυτή είναι μια μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αντιμετωπολίτευση οργάνωσε μια διαδήλωση η οποία κατεστάλλει διέως από τους πρετοριανούς του Προέδρου. Πολλοί άνθρωποι ε, σκοτώθηκαν, κακοποιήθηκαν, πολλές γυναίκες ευιάστησαν και εξεχιλιάστησαν επιπλέον. Ζητούμε λοιπόν να υπάρξει η διακοπή, η αναστολή της συμφωνίας αλίας με την χώρα αυτή. Και ζητούμε επίσης από την Αφρικανική Ένωση να επιβάλλει κυρώσει σε αυτή τη στρατιωτική χούντα και να κάνει προσπάθειες να υπάρξει συμφιλίωση και μια μεταβατική κυβέρνηση για να προετοιμάσει προεδρικές και βουλευτικές εκλογές και να θέσει στο περιθώριο αυτή τη χούντα που είναι εκτός της διεθνούς νομιμότητας. Αυτό είναι η απαραίτητη αντίδραση στο μεγάλο δράμα το οποίο έλαβε χώρα στη Γουινέα για να τονίσουμε επίσης με αυτόν τον τρόπο ότι και σε άλλες περιπτώσεις κατάφορης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει το θάρρος να δράσει με την ίδια οκίτητα και αποφασιστικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντοκεζέ. Η κυρία Βέμπερ για δύο λεπτά παρακαλώ. I'm Συγγνώμη, δεν άκουσα το όνομά μου. Εξετάζοντας την κατάσταση στη Γουινέα, και μαθαίνοντα για τι βιότητε που έχουν λάβει η χώρα του τελευταίου μήνε, το πρώτο θέμα που πρέπει ευλόγω να, να, να, να, αναφέρουμε είναι πώ δεν έχει καλυφθεί επαρκώ από τα μέσα α, αυτή η κατάσταση. Γιατί εκατοντάδες ε, θάνατοι, βασανιστήρια, αναξιοπρεπείς πράξεις έχουν λάβει χώρα. Οι διεθνή, τα διεθνή όργανα έχουν καταδικάσει την Χούντα που ανέλαβε την εξουσία μετά το πραξικόπημα, αλλά θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ περισσότερα για την βελτίωση της συνειδητοποίησης από πλευρά του κοινού, της κοινής νόμης και ιδιαίτερα των Ευρωπαίων πολιτών. Χαίρομαι που τουλάχιστον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιλώντας με τη φωνή των πολιτών, αναλαμβάνει δράση. Το ψήφισμα που θα ψηφίσουμε σήμερα δίνει μια απάντηση. Πλην όμως, το πιο σημαντικό είναι όχι μόνο να επικρίνουμε και να καταδικάσουμε το καθεστώς, αλλά και να αποφύγουμε κοινοτικοί πόροι να χρησιμοποιηθούν εναντίον των πολιτών της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέμπερ. Επόμενος ο κύριος Πρέντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 28 Σεπτεμβρίου, που είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία για το λαό της Γουινέας Κονακρή, ήταν ακριβώς η ημερομηνία του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία αυτής της χώρας. Αλλά από εφέτος θα είναι μια μαύρη ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου γιατί θα είναι και το σύμβολο της τρομερής σφαγής που οργάνωσε η στρατιωτική κυβέρνηση στην Γουινέα Κονακρή. Ήταν μια σφαγή κατά της αντιπολίτευσης στη χώρα αυτή. Με στόχο τη διατήρηση των στρατιωτικών στην εξουσία, κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχτεί. Ο λοχαγός Δαντής Καμάρα είχε είχε υποσχεθεί να εγκαταλείψει την εξουσία και να μείνει υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές. Τώρα που έχει εκπνεύσει το τελεσίγραφο της ε, Οργάνωσης για την Αφρικανική Ενότητα, είναι σαφέ ότι δεν μπορούν να παραμείνουν στρατιωτικοί στην εξουσία. Πρέπει να ασκήσει η διεθνή κοινότητα πίεση για εκλογέ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φρέντα. Για δύο λεπτά ο κύριο Βεζιά έχει το λόγο. Η κυρία Βεζιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω εκφράσει την άποψή μου ήδη στις Βρυξέλλες στην Μίνη Ολομέλεια πριν από 15 μέρες για το θέμα αυτό. Δεν θα επανέλθω σε αυτά τα οποία είπα τότε. Οι συναδελφοί μου γνωρίζουν ήδη και έχουν εκφράσει πάρα πολλά από τα πραγματικά γεγονότα. Εγώ νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει όλες οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ανταποκριθούν στην έκκληση που έχει κάνει η κοινωνία των πολιτών στη Γουινέα Κόνακρη για να φύγουν από την εξουσία οι στρατιωτικοί και οι οποίοι έχουν καταστήλει με πολύ βίαιο τρόπο την διαδήλωση η οποία έλαβε χώρα στις 28 Σεπτεμβρίου επέτειο της ανεξαρτησίας της Γουινέας. Μας ζητά η κοινωνία των πολιτών να βοηθήσουμε και θα ήταν πραγματικά απολύτως απαράδεκτο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγνοήσει αυτό το, αυτή την έκκληση και να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την αλληλευτική συμφωνία με τη Γουινέα Κονακρή, χρήματα που ξέρουμε θα πάνε κατευθείαν στα θυλάκια των στρατιωτικών και δεν θα πάνε για να βοηθήσουν τους αλληλείς της Γουινέας όπως προβλέπεται από την συμφωνία μας. Το καθεστώς είναι ένα αιμοσταγές, ένα διεφθαρμένο, στο πιο διεφθαρμένο καθεστώς στον κόσμο, δεν το λέω εγώ, το λένε οι φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν η θερμή μου παράκληση όλοι να ψηφίσουμε το σύνολο του κοινού ψηφίσματος με όλες τις παραγράφους που ζητούν την αναστολή της αλληλευτικής συμφωνίας με τη Γουινέα Κονακρή και ελπίζω ότι εδώ θα μας ακολουθήσει και το Συμβούλιο καθώς και η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Μπιλάν ένα λεπτό. Πρόεδρε, στο τέλος του περασμένου έτους, μετά το θάνατο του πρόεδρου Κόντε, ο λοχαγός Καμάρα ανέλαβε την εξουσία στη Γουινέα. Τότε πιστέψαμε, τον πιστέψαμε όταν είπε ότι θα προκηρύξει ελεύθερες εκλογές και δεν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος. Σήμερα κατανοούμε ότι κάναμε λάθος πάνω από 50.000 άτομα στις 28 Σεπτεμβρίου 2008 μαζεύτηκαν στο κεντρικό στάδιο για να διαμαρτυρηθούν ε, εναντίον του λοχαγού. Του συνάντησε ο θάνατος δυστυχώς. Στρατιώτες σκότωσαν περίπου 200 άτομα, ε, βίασαν πολλές γυναίκες, τραυμάτισαν χιλιάδες ανθρώπους. Ο κύριος Σολάν αντέδρασε ταχύτατα και εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του στην ε, γαλλική κυβέρνηση που απέφυγε να συνεργαστεί με τις αρχές Γουινέας. Πλην όμως, τρεις βδομάδες μετά από, αυτή την καταστροφή, από αυτές τις φαγές, ε, δεν βλέπουμε να ασκείται άλλη πίεση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται κυρώσει όσο πιο αυστηρέ γίνεται. Γιατί μόνον έτσι μπορούμε να αναμένουμε ότι ο Λοχαό Καμάρα θα εγκαταλείψει την εξουσία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφαση την οποία έλαβε, την απόφαση του Επιτρόπου Τζο Μπόρτς, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα, λέγοντας ότι η Κομισιόν αποσύρει την πρότασή της για μια αλληλευτική συμφωνία με τη Γουινέα. Ήδη έχει πει όχι σε αυτή τη συμφωνία μετά, δύο μέρες μετά από την σφαγή, όπου πάνω από 150 άτομα πυροβολήθηκαν από τις κυβερνητικές δυνάμεις που ελέγχονται από τον λοχαγό Καμάρα. Ελπίζουμε ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για αναστολή λοιπόν της Αλληλευτικής Συμφωνίας και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναθεωρήσει πλήρως την εμπορική της πολιτική έναντι των απθεσιωμένων χωρών φέρουμε βαριά ευθύνη για τα θέματα αυτά, γιατί είμαστε μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εμπορικές δυνάμεις. Σίγουρα σε σχέση με τους εταίρους της Αφρικής και επίσης ένας από τους μεγαλύτερους φορείς σε σχέση με την ανάπτυξη. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τη σχέση εμπορίου και ανάπτυξης και φυσικά και τη σχέση που διατηρούμε με ένα τέτοιο καθεστώς. Η αληθική συμφωνία με τη Γουινέα Κονακρή είχε σαν στόχο να βελτιώσει την κατάσταση Πέραν των χρηματοδοτήσεων, λοιπόν, για την ε, βελτίωση της αλληλείας, είχε σαν στόχο να βελτιώσει το γενικό βιωτικό επίπεδο. Φαίνεται όμως, ότι τα χρήματα αυτά αυτή τη στιγμή πηγαίνουν να υποστηρίξουν κατευθείαν το στρατιωτικό καθεστώς, κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθούν οι ομιλητέ εξ ονόμαστε των πολιτικών ομάδων. Ο κ. Κάτσμαρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πριν από δύο εβδομάδες μίλησαν ξανά για την Γουινέα. Δυστυχώς η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί την προσοχή μας και την αντίδρασή μας. Τη Δευτέρα η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, είδε την δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού κ. Διάλο που ήταν αυτόπτης μάρτυρας των επεισοδίων της 28 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι αρκετό να ζητούμε, ή να απαιτούμε η Χούντα να ε, σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο, το, αν το στρατιωτικό καθεστώς σεβόταν τέτοιου είδους δικαιώματα δεν θα θεωρεί το στρατιωτικό καθεστώς. Χρειάζεται πράξεις και όχι μόνο λόγια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάτσμαρεκ. Ε, ο κύριος ε, Τυρολιάν διορθώνει ο πρόεδρος. Η Γουινέα τραντάζεται από δραματικά γεγονότα που έχουν εκπλήξει την κοινή γνώμη και έχουν παραβιάσει τον δρόμο. από τις 28 Σεπτεμβρίου η Χόντα του κ. Καμαρά ε, έπνιξε στο αίμα την ε, διαδήλωση εναντίον της. Όμως οι συμφωνίες του Κοτονού αποτελούν θεμέλιο τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και απαιτούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών τη δημοκρατία. Αν ο λοχαγός ε, Καμαρά αποφάσισε μόνο μερός να αναβάλει τις εκλογές και να καταπνίξει τις ε, διαδηλώσεις, αυτό αποτελεί σημαντική παραβίαση τη θέση που είχε αναλάβει να διοργανώσει εκλογέ σε ένα χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσει σύμφωνα με τι αρχέ και τι πάγιε αρχέ ε, που την χαρακτηρίζουν, έτσι ώστε να σταματήσουν τα βία επεισόδια που αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαίρομαι, συμβαστικό ψήφισμα συνάδει με τις αρχές μας και τις αξίες μας. Όμως, θέλω να επιμείνω στο άρθρο 10 την αναστολή του πρωτοκόλου ε, αλληλευτικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία της Γουινέας. Όσο η δημοκρατική διαδικασία δεν ε, εξελιχθεί, δεν ξεκινήσει, θα πρέπει να, ανασ... να παραμείνει υπό αναστολή. Η... Ε, θα έχει ασφαλώς αυτή η αναστολή αποτελέσματα επί του πληθυσμού, πλην όμως έτσι κι αλλιώ, τα αιματηρά επεισόδια τη 28 Οκτωβρίου καταδίκασαν τον πληθυσμό σε εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση. Από το 1968, από την ανεξαρτησία, η Γουινέα έχει γνωρίσει μόνο δικτατορίε. Ευχαριστώ κύριε Τυρολιά. Ο κύριο Χάγλουντ, επόμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα εγώ να επαναλάβω αυτό που είπαν οι προαλήσαντες συνάδελφοι. Θα ήθελα όμως να τονίσω ξανά ότι χαίρομαι που ξανασυζητούμε αυτό το θέμα σήμερα εδώ. Στην Επιτροπή Αλίας το συζητήσαμε στις 30 Σεπτεμβρίου. Γιατί μας απασχολεί αυτό το θέμα. Κανονικά θα έπρεπε να διακοπούν όλες οι ελευτικές συμφωνίες. Και όχι μόνο οι ελευτικές και όλες οι εμπορικές συμφωνίες. Είναι πραγματικά αξιοθρήνητη η κατάσταση και το ψήφισμα τα περιγράφει πολύ καλά. Το ζήτημα της αλίας είναι ένα και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι άλλο. Να δούμε πώς αντιδρούν οι πολιτικοί. Στην Επιτροπή Αλίας θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν οι εμπορικές συμφωνίες και η ελευτική συμφωνία με χώρες όπως η Γουινέα. Είναι σχετικά λοιπόν ε, μεγάλη συμφωνία, για να μην πω ομόφωνα, συμφωνεί Επιτροπή Αλίας πλέον να ε, διακοπεί, να ανασταλεί η συμφωνία. Τελικά καταλήγω ότι είναι θετικό αυτό. Μπορεί να θεωρήσετε ότι τα όσα έγιναν στη χώρα έπληξαν και την αλία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια αηφόρο κατάσταση, μια αηφόρο συνεργασία και μόνιμη και σταθερή. Διότι χρειάζονται εισόδημα και οι άλλοι, Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζωμέβα Ιρουέντα. Συμμετείχα στην, Επιτροπή, στην ε, συνέδρια της Επιτροπής Αλίας όταν ψήφισε με μικρή βέβαια διαφορά αλλά υπερψήφισε τη μία ε, ανανέωση συμφωνίας Αλίας εξαιτίας ε, των, της των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των σφαγών κλπ. της αιματοχυσίας που ε, ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί και δεν έχουν διαρευνηθεί. Θα ήθελα η Ολομέλεια να επιβεβαιώσει αυτή την απόφαση Επιτροπή Αλία. Γιατί έτσι θα στέλναμε μια, ένα σαφέ μήνυμα και στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κυβέρνηση τη Γουινέα ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι με χρήματα των πολιτών μα να συνεισφέρουμε στο να διατηρηθεί στην εξουσία μια τέτοια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Για μια φορά τουλάχιστον χαίρομαι και ελπίζω να αποτελέσει προηγούμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ανθρώπινε ζωέ δείχνουν να είναι πιο σημαντικέ από μια απόφαση πολιτική σημασία, από μια συμφωνία πολιτική σημασία. Η Επιτροπή Αλία το ψήφισε. Θα πρέπει και η Ολομέλεια να επιβεβαιώσει αυτή την απόφαση. Είναι μεγάλη ευκαιρία που ανοίγεται μπροστά μας και ελπίζω να διατηρηθεί και το άρθρο 10 όπως έχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρομεδά Ιρουέδα. Τέλος από τις πολιτικές ομάδες ο κύριος Πορέβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τουλάχιστον 157 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.200 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της ειρηνικής διαδήλωσης της ε, αντιπολίτευσης σε ένα μεγάλο στάδιο στο Κονακρή αυτό την επέτειο της ε, ανεξαρτησίας της Γουινέας Κονακρή το 1968. Όταν ο Λοχαγός Καμάρα πήρε την εξουσία πέρσι το Δεκέμβριο, είχε υποσχεθεί να ξαναδώσει την εξουσία σε πολιτική εξουσία μετά από δημοκρατικές ε, εκλογές. Δεν έχει τηρήσει την υποσχεσή του, αξακολουθεί να είναι μια στρατιωτική χούντα η οποία κυριαρχεί στη χώρα αυτή με απόλυτη περιφρόνηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουν σκοτώσει, έχουν τραυματίσει, έχουν διάσει. Ω εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εμεί θα πρέπει να εγείρουμε το ανάστημά μα για να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου, να εξασφαλίσουμε ότι η Χούντα θα τιμωρηθεί και ότι αυτέ οι ομότητε δεν μπορούν να συνεχιστούν. Η Γουινέα είναι μια χώρα τεράστιου οικονομικού δυναμικού, αλλά εξακολουθεί να είναι μια από τι φτωχότερε και πιο διεφθαρμένε χώρε στην Αφρική οποιαδήποτε συνέχιση της στρατιωτικής χούντας μπορεί να οδηγήσει σε ένα εμφύλιο πόλεμο και σε γενικότερη ανάφλεξη της περιοχής της Δυτικής Αφρικής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πορέβα. Η κυρία Ντελβό, για ένα λεπτό. 157 νεκροί και πόσες σεξουαλικές ταπεινώσεις στις 28 Σεπτεμβρίου, μια χωρίς προηγούμενο βία που εξαπολύθηκε κατά του λαού της Βοηνέας Κονακρή. Είναι μια αντίδραση δυσανάλογη ακόμα και από μια στρατιωτική χούντα και ενώπιον αυτής της βαρβαρότητας εμείς θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα στεναροί. Εγώ χαίρομαι για τις στοχευμένες κυρώσει που αποφασίστηκαν από τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον του καθεστώτο Καμάρα. Ενώπιον αυτών των γεγονότων δεν αρκεί βέβαια κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρξει άπλετο φω σε σχέση με τα γεγονότα από μια πραγματικά διεθνή επιτροπή έρευνα και τα εγκλήματα αυτά δεν πρέπει να μείνουν στα επίπεδα ατιμορρεσία. Είναι απαραίτητο επίση να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα στη διάθεσή τη για να μπορέσει να δράσει κατά, τον, κατά τη σεξουαλική βία σαν όπλο πολέμου. Κάτι το οποίο συμβαίνει σε πολλέ περιοχέ ένοπλων συγκρούσεων. Πολλέ φορέ είναι οι πολύ νέε, οι πολύ ηλικιωμένε γυναίκε οι οποίε θίγονται, εν πάση περιπτώσει, τα πιο ευαίσθητα και τροτά άτομα. Εμεί θα πρέπει να ζητήσουμε το κράτο του δικαίου, την καλή διακυβέρνηση αλλά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία των πιο τροτών τμήματων του πληθυσμού σαν απαράγραπτη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία συνεργασίας στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντελβό. Και τώρα κύριος Δεζίερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, 28 Σεπτεμβρίου ο λαός της Γουινέας ε, διαδήλωνε για να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις για ελεύθερες εκλογές δημοκρατικές και έπεσε θύμα της χείρισης καταστολής από ένα καθεστώς που στερεί το κάθε νομιμότητας και εκείνη τη μέρα έχασε οποιαδήποτε αξιοπρέπεια του είχε απομείνει ξεκύλιαζαν γυναίκες με μπαγιονέτες, τις βίαζαν, ε, ε, βασάνιζαν ε, αντιφρονούντες και συνδικαλιστές της αντιπολίτευσης. Εμείς θα πρέπει να είμαστε στο πλευρό της Αφρικανικής Ένωσης και των άλλων διεθνών οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών για να μην αφήσουμε τιμότητα αυτά τα εγκλήματα και πάντα στο πλευρό του λαού της Γουινέας. Είναι μια χώρα που βρήθη πλούτου, δεν θα μπορέσει ποτέ να αναπτυχθεί εάν δεν ξεφορτωθεί τους δικτάτορες και ε, τις κλίκες που κυβερνούν. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα συζητούμε αυτό. Δεν μπορούμε όμως από τη μια να βλέπουμε το στενό οικονομικό συμφέρον και από την άλλη τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει όσοι έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Κοτομού νου, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και οφείλουμε στο λαό της Γουινέας να είμαστε στο πλευρό του, στον αγώνα του για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεζίρ. Ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία κατς the Ο κύριος Κατσουλίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο για να κάνω ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά την πρόταση αναστολής της ε, ε, αληφτικής, του αλληλευτικού πρωτοκόλλου Ευρωπαϊκής Ένωσης Γουινέας. Ε, αμφιβάλλω για το κατά πόσον ε, ένα βάναυσο καθεστώς ε, που θυσιάζει 156 ζωές από τους πολιτών του θα συγκινηθεί από μια τέτοια δυσανάλογα μικρή ποινή κύρωση. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για νομικές υποχρεώσεις έναντι των πολιτών αυτής της ε, χώρας που δεν έχουν καμία σχέση με το καθεστώς και ασχολούνται με τον τομέα της αλίας. Γι' αυτό το λόγο το ΕΛΚ διστάζει σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κασουλίδη. Ο κύριος Τάνοκ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ιστορία της Γουινέας Κονακρή ακολουθεί ένα απόλυτα απογοητευτικό αφρικανικό σενάριο. Δικτατορίες, στρατοδιωτικά καθεστώτα, εναλλαγή δικτατορικών και αυταρχικών καθεστώτων που αφήνουν το λαό του σε απόλυτη ένδια. Οι ορυκτή πόροι θα μπορούσε να κάνουν τη Γουινέα ένα από τα πιο ευμαρή αφρικανικά κράτη. Αντίθετα όμως ο λαός της ζει σε απόλυτη αθλειότητα. Και η Γουινέα όπως και όλη η περιοχή έχουν γνωρίσει μονάχα αιματοχυσία και αστάθεια τα τελευταία 20 χρόνια. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει μια διαδικασία Κίμπερλε όχι μονάχα για τα διαμάντια αλλά και για άλλα ορυκτά ώστε οι εξορυκτικές εταιρείε να μην υποστηρίζουν τους εμφύλους πολέμους ή αιμοσταγή καθεστώτα όπως αυτά του Καμάρα. Και επίσης υπάρχουν πολλές συμφωνίες μεταξύ της Γουινέας και των κινέζικων εταιριών. Ελπίζω ότι η Κομισιόν θα εκφράσει προς το Πεκίνο την άποψή της ότι αυτές οι εμπορικές συμφωνίες δεν πρέπει να υποστηρίξουν εμφύλιο πόλεμο και περαιτέρω αιματοχυσία στο, στην Γουινέα. Συμφωνώ με τον κύριο Κασουλίδη ότι μια αναστολή της αλληλευτικής συμφωνίας θα πλήξει το λαό και όχι το στρατιωτικό καθεστώς. Ευχαριστώ κύριε Ταν Νοκ. Η κυρία Χάουταλα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα, που όλοι έχουν εκφράσει την ευγνωμοσύνη τους προς την Κομισιόν για την απόφαση που ελήφθη σε σχέση με την Αλληλευτική συμφωνία λόγω της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Επίτροπο αν η δική σας πρόθεση είναι να προχωρήσετε με τρόπο συστηματικό να αναλύσετε παρόμοιες καταστάσεις ώστε να έχουμε μια συνεκτικότητα στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τέτοιου είδους εμπορικές συμφωνίες όταν ανακύπτουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Ευχαριστώ. Η κυρία Κορχολά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, ένας ε, Δανός πιοφόρος με ρώτησε πώς μπορούμε να ορίσουμε την έννοια ανθρώπινα δικαιώματα και του απάντησα εγώ δεν χρειάζεται να ορίσω αυτή την έννοια δεν θα είχε νόημα να την, να την ορίσω εγώ ίδια. Ο ορισμός αυτός ήδη υπάρχει. Και, όποιοι, και τα κράτη, όλα τα κράτη είναι υποχρεωμένα να σέβονται αυτόν τον ορισμό και να σέβονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Γουινέα έχει συνυπογράψει τη Συμφωνία Κοτονού, σύμφωνα με την οποία είναι υποχρεωμένη να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η κίνηση, αυτή είναι η αφετηρία και οποιασδήποτε άλλε συμφωνίε βασίζονται στη συμφωνία στο πρωτόκολλο του Κοτονού, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτή την πραγματικότητα. Θα πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα και ενδεχομένω να επιβάλλουμε και κυρώσει. Υπάρχουν πολλά μεταλλεύματα, σύνδρομα μεταλλεύματα στην ε, Γουινέα. Είναι ένα από τα πιο διεφθαρμένα καθεστώτα. Είναι πολύ κρίμα που κινέζικες εταιρείε επενδύουν στην Γουινέα και, δεν απαιτούν κανένα ε, είδους προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Καθεστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει μετά το τέλος της συζήτηση για τα κατεπήγον. Um Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, αλλήμον ξέχασα τον Επίτροπο. Παρακαλώ, κύριε Όρμπαν. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, γρήγορα και με στένος καταδίκασε Μπορώ να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ζήτησε κάποιο το λόγο για διαδικαστικό. Τι θέλετε για διαδικαστικό, ζητήσατε το λόγο, αγαπητέ συνάδελφε. Όχι, όχι. Στο Catch Ναι, λυπάμαι πάρα πολύ, αγαπητέ συνάδελφοι. Είχαμε προβλέψει δύο λεπτά, έδωσα το λόγο σε τέσσερι συναδέλφου, δύο από το ΕΛΚ. Τι να κάνουμε, τώρα πρέπει να μιλήσει ο Επίτροπο. Παρακαλώ, κύριε Όρμπαν. Comisia Έλεγα λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα και στεναρά καταδίκασε ε, την αιματοχυσία και το μακελιό και την παραπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 28 Σεπτεμβρίου του 2009 που συνεχίστηκαν και τις επόμενες ημέρες. Συμμετέχοντας στη Διεθνή Επιτροπή για στη Γουινέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα συμπεράσματα της 12ης ε, Οκτωβρίου που προβλέπουν πολλά μέτρα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταρχάς, από ανθρωπιστική σκοπιά θα πρέπει όσοι κρατούνται αυθαίρετα να απελευθερωθούν. Επίσης, οι σωροί των θυμάτων να επιστραφούν στις οικογένειες και ε, οι τραυματίες, κυρίως οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμού, να ε, τύχουν της απαραίτητης ιατρικής ε, περίθαλψης. Εκφράζουμε τη λύπη μας και την ανησυχία μας, διότι από ό,τι φαίνεται προς το παρόν κανένα από τα μέτρα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί. Δεν έχει εφαρμοστεί, συγγνώμη. Ε, στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να συγκληθεί Διεθνής Επιτροπή ε, Διερευνητική που θα εξετάσει ε, τα ε, γεγονότα της 28 Σεπτεμβρίου και τη δηματοχυσία για να έρθουν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα πρέπει να τερματιστούν αυτές οι καταστάσεις στη Γουινέα. Η Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή θα κάνει μια προκαταρκτική έρευνα και εξέταση ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και Πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει να βελτιωθεί η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να αναλύσει τη δυνατότητα ή το ενδεχόμενο οικονομικής στήριξης για μια διεθνή αποστολή παρατήρησης και προστασίας, έτσι ώστε να υπάρχει προστασία των μελών και των μαρτύρων, για να μην έχουμε φαινόμενα εκφοβισμού και να επικρατεί στη χώρα ασφάλεια. Εκτός από πλήρη απαγόρευση εμπορίου ε, όπλων, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προτείνει μέτρα για την ασφάλεια, για μεταρρύθμιση των όπλων δυνάμεων, έτσι ώστε η χώρα αυτή να ανακτήσει την ασφάλειά της. Τέλος, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι τα μέτρα που εδώ επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού έχουν ληφθεί ήδη από τις 27 Ιουνίου. Και για λόγους συνέπειας συνέχεια για να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή στη στρατιωτική χούντα, ο ο αρμόδιος επίτροπος ο κύριος Μπόρτς ανακοίνωσε ήδη την πρόθεσή του να αποσύρει την πρόταση συνεργασίας ε, και της αλληλευτικής συμφωνίας που ε, πρόκειται να συναυθεί με τη Γουίνε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρξει καμία πληρωμή σχετική με το πρωτόκολλο αυτό. Και για να απαντήσω και στην ερώτηση που μου κάνατε, είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λαμβάνει ε, μέτρα αναλύοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά και κάθε κατάσταση ξεχωριστά, βλέποντας και κάνοντας. Ευχαριστώ κύριε Όρμπαν. Ε, τώρα ολοκληρώνει τη συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει μετά το τέλος της συζήτησης για τα κατεπήγοντα. Ακολουθεί τώρα η συζήτηση για 7 προτάσεις ψηφίσματος για το Ιράν. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους συντάκτες. Η κυρία Γκόμες.